Έχουμε λάβει μια αίτηση του ΕΛΚ για την αντικατάσταση της κυρίας Σουίτς την προσωπία με την Ουκρανία. Υπάρχουν σχόλια σχετικά. Εγκρίνεται αυτή η αλλαγή. Έχουμε λάβει την θέση σε πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου